όταν αυτό ε, δια νόμου απαγορεύεται. Αλλιώ είναι δημαγωγία και λαϊκισμό. Κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, έληξε η συζήτηση εδώ και η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο στι 12. Τώρα ερχόμαστε στο επόμενο θέμα της ε, ημερήσιας διάταξης. Είναι η έκθεση του κυρίου Ιβάν «Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης κατά πολέμηση της απάτης» Θα αρχίσουμε τη συζήτησή μας με τον εισηγητή. Κύριε Ιβάν, έχετε το λόγο για τέσσερα λεπτά. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, η έκθεση αυτή αφορά την προστασία των οικονομικών συμφετάρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βασίζεται σε μια ανακοίνωση της Επιτροπής ε, βάσει του άρθρου 139 της Συνθήκης. Εκεί γίνεται σαφής αναφορά στην καταπολέμηση της απάτης. Ε, η ανακοίνωση της Επιτροπής όμως δεν αναφέρεται σαφώς, ε, με, αναφέρεται σαφώς ποιες θεωρούνται απάτες και ποιες θεωρούνται απλά λάθη. και επίσης δεν ξεχωρίζεται η συμπεριφορά η οποία είναι πραγματική διαφθορά ή η συμπεριφορά η οποία απορρέει από ενδεχόμενα λάθη. Ε, υπάρχει επίσης μια ανοχή για τα λάθη αλλά ε, και αν υπάρχει μια τέτοια ανοχή δεν είναι δυνατόν να υπάρξει και για την απάτη. Η απάτη για την απάτη η ανοχή είναι μηδενική, κυρίως όταν μιλάμε για τον προϋπολογισμό της Ένωσης. Ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα είναι αυτό το οποίο συνδέεται με την συλλογή πληροφοριών και δεδομένων. Πρέπει να μιλήσουμε πολύ σοβαρά για τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη-μέλη ε, μεταδίδουν ε, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πληροφορίες ε, σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούν το ευρωπαϊκό χρήμα, τους ευρωπαϊκούς πόρους. Οι εκθέσεις ε, τις οποίες διαβιβάζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι ε, σαφώς υψηλότερης ποιότητας. Ρώτησα τον ε, Επίτροπο ε, έτσι ώστε να μου πει αν είναι δυνατόν οι δηλώσεις των κρατών μελών να υπογράφονται είτε από τον Υπουργό ε, Οικονομικών είτε από τον επικεφαλής της ε, κυβέρνησης. Κάτι τέτοιο θα ήταν δεσμευτικό για τα κράτη. Είναι πάρα, πολλά, πάρα πολλοί οι πόροι οι οποίοι χρησιμοποιούνται και οι οποίοι προέρχονται ε, κυρίως από, το, από τους ε, δασμούς. 70% των πόρων ε, διέρχονται μέσω απλουστευμένης διαδικασίας. Από το 2001 μέχρι το 2010 έχει καταδειχθεί ότι ο έλεγχος για την απλουστευμένη διαδικασία είναι πάρα πολύ χαμηλός και ότι τα ποσοστά λαθών είναι εξαιρετικά ψηλά πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υπάρξει μελέτη σχετικά με τον αντίκτυπο των λαθών αυτών. Θα ήθελα εδώ να συγχαρώ την Όλαφ ε, για την επιχείρηση Διάβολο 2 που όχι μόνο στοχεύει στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, αλλά θέλει να καταπολεμήσει και την ε, παραχάραξη. τα προϊόντα απομίμησης ε, προκαλούν πάρα πολύ μεγάλη καταστροφή αλλά από την άλλη πλευρά δεν μιλάμε μονάχα για απώλεια χρημάτων μιλάμε και για απώλεια της εμπιστοσύνης των πολιτών. Η χρήση των πόρων ε, βεβαίως γίνεται λόγος ε, από την μία πλευρά ε, για την σωστή χρήση των πόρων ενώ από την άλλη μεριά πρέπει να δούμε τι γίνεται με τους πόρους που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί. Το σύστημα οικονομικού ελέγχου σε αυτή την περίπτωση μπορεί να είναι καλό όμως αντιμετωπίζει πολύ μεγάλες δυσκολίες γιατί βασίζεται σε στοιχεία και σε βάσεις δεδομένων που παρουσιάζουν πολλά λάθη την ίδια στιγμή εάν ε, μιλάμε για ανάκτηση των ευρωπαϊκών ε, πόρων πρέπει να πούμε ότι ε, έχουμε 32% των πόρων που προέρχονται χρησιμοποιούνται στη γεωργία και φτάνουμε σε πολύ ψηλότερα ποσοστά όταν μιλάμε για τα διορθωτικά ταμεία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σιγητά. Το λόγο θα πάρει ο Επίτροπος ο κύριος Σεμέτα. You have the floor, Commissioner. Uh, Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τον εισηγητή, τον κύριο Ιβάν, για μια πολύ επικοδομητική γνωμοδότηση και θα εστιάσω την παρέμβασή μου σε έξι κομβικά σημεία. Για τις πληροφορίες που παρέχονται από την έκθεση για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων. Στην έκθεση του 9 ήδη ε, δίναμε λεπτομερείς πληροφορίες για τα επίπεδα παρατυπιών και απάτης που είχαν διαπιστωθεί ανά μέλος για την περίοδο 2006 συνοχή. Λαμβάνω βέβαια υπόψη τις προτάσεις σας και τις καταγράφω. Δεύτερον, για την συνθήκη για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων προετοιμάζω μια ανακοίνωση που θα παρουσιαστεί με την Αντιπρόεδρο κυρία Ρέντινγκ τον Μάιο για την προστασία των δημόσιων κονδυλίων από όλων των ειδών της παράτυπες συμπεριφορές όπως την απάτη, τη δωροδοκία και όλα αυτά για να αποκτήσουμε ένα νέο νομικό πλαίσιο. Για τους ίδιους πόρους, το 2010 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άρχισε ε, να επισκέπτεται όλα τα κρατημέλη για να διαπιστώσει πώς λειτουργούν αυτές οι απλουστευμένες τελωνιακές διαδικασίες. Και όλα αυτά θα παρουσιαστούν ε, αφού αναλυθούν σε μια έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όπου θα εξετάζουμε επιδόσεις ε, και σφάλματα τα τσιγάρα έχουμε συνάψει συμφωνίες με τέσσερις καπνοβιομηχανίες και θα συνεχίσουμε να πιέζουμε προς την ε, σύσταση και υποθήκης για τον έλεγχο των λαθρέων προϊόντων καπνού. Ελπίζουμε κάτι παρόμοιο με αυτό που έχει υπογραφεί σε επίπεδο ΠΟΗ. Βεβαίως έχουμε και το πρόβλημα των απατών και των παρατυπιών που ε, διαπιστώνουμε στην ε, ΚΑΠ και έχουμε ε, καταλογισμούς που φτάνουν το 10% σε αιτήσιο επίπεδο ανάλογα με τη σοβαρότητα της παρατυπίας. Για το 2012 προτείνουμε μια απλούστευση και αν θέλετε, διευκόλυνση της διαδικασίας για τις δημόσιες συμβάσεις για να λάβουμε υπόψη όλες αυτές τις παραμέτρους. Η διαδικασία για την ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών αποτελούν και μια εξασφάλιση ότι η διαδικασία λειτουργεί σωστά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρησιμοποιεί την διακοπή και αναστολή πληρωμών πολλές φορές ε, για να συνετίσει κράτη-μέλη όπου τα συστήματα ελέγχου και παρακολούθησης χρήσης κοινοτικών και ενδολίων δεν είναι Είχαμε 4 δις εκατομμύρια ευρώ πληρωμών στο χώρο της συνοχής και των διορθωτικών ταμείων που ανεστάλησαν την περασμένη χρονιά. Και για την ανάκτηση από τον τελικό, ε, από τον τελικό δικαιούχο υπεύθυνα πάντα είναι ε, τα κράτη-μέλη. Για την Γεωργία η ανάκτηση έφτασε τα το 33% για υποθέσεις το 2007, μια βελτίωση δηλαδή με το 10% που έχουμε για τις υποθέσεις οι οποίες χρονολογούνται από πριν το 2006. Για τα πολυετή προγράμματα βεβαίως η πλήρης εικόνα ε, θα διαπιστωθεί πώς έχει αφού λήξει η περίοδος εκταμίευσης ε, και βέβαια θα πρέπει να αξιολογηθούν και οι επιδόσεις των κρατών μελών να βρούμε αν είναι ικανοποιητικέ ή όχι. Εμείς κάνουμε ένα follow-up ε, σύμφωνα με τις προτάσεις του Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Κύριε Επίτροπε, τώρα το λόγο θα πάρουν ομιλητέ εξ ονόματος των πολιτικών ομάδων για την ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος η κυρία Μακόβε για δύο λεπτά παρακαλώ. Um, Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι θα πρέπει να μιλήσουμε για ε, τα σημεία τα οποία πρέπει να διορθωθούν. Άρα τα κρίσιμα σημεία. Πρώτο μεταξύ αυτών αναφέρεται στο γεγονός ότι η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν δίνει πληροφορίες σχετικά με το ποσοστό παρατυπιών, αν παρατυπιών ε, ανακράτος. Αυτό θα μας επέτρεπε να έχουμε ε, μια καλή αναλυτική εικόνα για τις παρατυπίες και τις απάτες της χώρας. Επίσης, ε, ασχολείται ευρέως με τις παρατυπίες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά δεν κάνει το ίδιο και με τις απάτες. Ελπίζουμε ότι του χρόνου θα το θέμα αυτό. Δεύτερον, δημόσιες ε, προμήθειες. Ε, αυτό είναι, είναι ένα πεδίο μεγάλης ε, διαφθοράς και πολλών παρατυπιών Ζητούμε από την Επιτροπή λοιπόν να εστιάσει στον, την προσοχή της στον κανονισμό των δημοσίων προμηθειών, να εφαρμόσει κατά αυτήν την έννοια ε, κοινέ ε, προϋποθέσεις, σαφείς ε, όρους και επίσης συγκεκριμένα κριτήρια βάσει των οποίων λαμβάνονται οι αποφάσεις και για τους δημόσιους διαγωνισμούς και επίσης να υπάρχει διαφάνεια όσον αφορά το, τους δημόσιους διαγωνισμούς. Ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο ε, να ε, ε, προχωρήσει στην ολοκλήρωση των διαδικασιών και μετά όσον αφορά τους δημόσιους διαγωνισμούς και επόμενο ζήτημα βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα όσον αφορά τους δικαιούχους των ευρωπαϊκών κονδυλίων στις χώρες μέλη. Θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει μία ενιαία ενιαία διαδικασία απλουστευμένη έτσι ώστε να μπορεί να υπάρξει έλεγχος ε, των ε, ε, διαδικασιών. Επίσης να υπάρχουν τυποποιημένες διαδικασίες ε, για όλους ε, και σε όλες τις περιπτώσεις ε, και μπορεί κανείς να διαβάσει πληροφορίες αυτές στην γλώσσα του γιατί διαφορετικά δεν θα υπάρχει διαφάνεια και θα μπερδευτούμε πάρα πολύ. Επίσης ο Επίτροπος μόλις είπε ότι πάντα υπάρχει δυνατότητα περαιτέρω βελτιώσεως. Την αναμένουμε λοιπόν τη βελτίωση αυτή. για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, αξιότιμη κύριε Επίτροπε, σε μετά. Γνωρίζουμε ότι το 80% των κονδυλίων της Ένωσης ε, είναι στη συνδιαχείριση, δηλαδή το διαχειρίζονται τα κράτη-μέλη και ε, τα δαπανούν. Και εκεί βλέπουμε τα σφάλματα, τις παρατυπίες, τις ατασταλίες και τις απάτες. Γι' αυτό η αιτήσια έκθεση για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι κάτι σαν το μητρό αμαρτιών ε, των κρατών μελών. Και ευχαριστώ και τον Κατλίν Σόριν και τους και ηγητές των άλλων πολιτικών ομάδων για το έργο τους. Έκθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Προστασία των Συμφερόντων Στη γερμανική εκδοσή σελίδα 11 λέει το εξής αξιοσημείωτο. Στα προγράμματα στόχου 2 ήταν μεγάλες παρατυπίες στις χώρες Ηνωμένο Βασίλειο και ε, ε, κάτω χώρες παρακαλώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, το Ηνωμένο Βασίλειο και οι κάτω χώρες είναι δύο χώρες που μας πρότειναν να μειώσουμε τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και δεν μπορώ παρά να καλέσω εδώ τις χώρες αυτές να πούνε με ασχοληθείτε με τη σωστή χρήση ε, των κονδυλίων των Ευρωπαίων πολιτών και μειώστε τις παρατυπίες και τις ατασταλίες σας. Αν έχετε να μας πείτε τίποτα κύριε Επίτροπε θα με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Στάς για την ομάδα των Πρασίνων για 1,5 λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι η καταγραφή ε, απατών και παρατυπιών ε, στην Ένωση είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον νομοθέτη. Μας δίνει πού πηγαίνουν τα χρήματα, ε, ποια είναι τα σφάλματα ενδεχομένως και πού χωράει βελτιώσει στο σύστημα. Εξού και η έκθεση είναι πάρα πολύ σημαντική. Μετά τη συζήτηση που είχαμε στην Επιτροπή Καταπολέμησης Απάτη στο Κοινοβούλιο μπορούμε να καταλήξουμε στα εξή. Πρώτον, οι εκθέσει θα πρέπει να είναι πιο συγκεκριμένε, πιο ακριβείς, να δοθεί προσοχή στην πραγματική ε, απάτη και στον πραγματικό όγκο παρατυπιών. Δεύτερον, τα κράτη-μέλη πρέπει να αναφέρουν καλύτερα. Ε, σήμερα δεν είναι βέλτιστη η κατάσταση, βέλτιστη και το λέω έτσι με μια ωραία κομψή έκφραση, αλλά θα πρέπει να πιέσουμε τα κράτη-μέλη ε, και να τα απειλήσουμε και με κυρώσεις. Τρίτον, τα χρεωστή τους καταβληθέντα ποσά θα πρέπει βεβαίως να επιστρέφονται και να ανακτώνται να πάρει τα κατάλληλα μέτρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα το συζητήσουμε και τον άλλο μήνα εδώ στο Στρασβούργο στη συζήτηση για την απαλλαγή. Εδώ έχω ε, ε, ε, να πω ότι είναι προβληματική η κατάσταση. Επίσης, θα πρέπει να δούμε πώς τα κράτη-μέλη διαπιστώνουν ε, τις απάτες. Η Ισπανία και η Γαλλία υπολείπονται. Εγώ είμαι μόνιμος συζητητής για τους ιδίους πόρους και θα ήθελα να ευχαριστήσω και να συγχαρώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κυρίως και την ε, Όλαφ για την καταπολέμηση των ε, απομιμήσεων τσιγάρων και προϊόντων καπνού. Είναι πραγματικά πολύ καλή η δράση αυτή που αναφέρθηκε διάβολο 2 και οι συζητήσεις και οι συμφωνίες που έγιναν με την British American Tobacco, με την Imperial Tobacco 500 εκατομμύρια ευρώ μας δίνει και μόνο. Αλλά αυτά τα χρήματα δεν θα πρέπει να χαθούν στο γορβανά των κρατών μελών. Θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν σωστά και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από τα κράτη-μέλη στην καταπολέμηση της απάτης, στην εφαρμογή και ενίσχυση των μέτρων αυτών στα κράτη-μέλη. Γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τα χρήματα που απέφερε αυτή η συμφωνία θα πρέπει να πιάσουν τόπο. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολύ. <clears throat> Σεβαστείτε το χρόνο σας παρακαλώ κύριε συνάδελφε. Ε, η κυρία Σέσκοβα για ένα λεπτό από τους ε, Ευρωπαίους Συντηρητικούς Μεταρρυθμιστές. Eh, Ευχαριστώ. Ε, υποδέχομαι και εγώ την έκθεση αυτή πολύ μεγάλη χαρά γιατί ζητάει μεγαλύτερη διαφάνεια στην καταπολέμηση της απάτης και αξίζει την υποστήριξή μας. Ήδη από πέρυσι συζητούμε για την ευθύνη των κρατών μελών ε, ως προς τον έλεγχο και την εκτέλεση των ε, κοινοτικών κονδυλίων. Είναι πολύ σημαντικό κάθε κράτος μέλος να προστατεύει τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να εξασφαλίζει τους απαραίτητους ελέγχους σε επίπεδο κράτους μέλους, ακριβώς για να προλαμβάνονται οι παρατυπίες και οι απάτες. Εδώ χρειάζεται λοιπόν καλύτερη και μεγαλύτερη συνεργασία κρατών μελών και Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, ε, για τη διαβίβαση των πληροφοριών. Και θα πρέπει να είναι πολύ αυστηρή η έλεγχη των εθνικών αρχών. Η σύμβαση για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων είναι άριστο μέσο. Η τσεχική δημοκρατία που αναφέρεται στην έκθεση αυτή δεν έχει κυρώσει μέχρι στιγμή τη συγκεκριμένη σύμβαση. θα πρέπει τα νομικά πρόσωπα να υφίστανται έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές και μάλιστα από τις διοκτικές αρχές, της δίωξη ποινικού δικαίου. Αλλά αυτό δεν το συζητάει καθόλου το Κοινοβούλιο στην Τσεχική Δημοκρατία. Επίσης θα ήθελα να αναφερθώ και πάλι σε ένα σημείο. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Ανδριάσεν έχει το λόγο από την Ευρώπη Ελευθερίας Δημοκρατίας για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε πρόβλημα πολύ συχνά με την διαφθορά ε, και την απάτη. όλα αυτά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από μια μηδενική ανοχή έχει μετακινηθεί προς ένα περιθώριο ε, ανοχής με ανάλυση κινδύνου. Νομίζω ότι αυτό χειροτερεύει την εντύπωση που δημιουργούμε και δεν βοηθάει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που προσπαθεί να πατάξει την δωροδοκία. Μόνο οι δύο των οποίων ανακοινώθηκαν τα ονόματα παρετήθηκαν. Πότε λοιπόν θα αναθεωρήσουμε την ομοθεσία για τους ευρωβουλευτές. Και κάποιος ευρωβουλευτής μάλιστα έφτασε σε σημείο να αρνηθεί στην Όλαφ το δικαίωμα έρευνας και ανάκρισης λέγοντας πως σε κάποιες χώρες δεν είναι ποινικό αυτό το αδίκημα και δεν θα ε, ερευνά το. Γιατί νομίζω πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να ζητάει από τα κράτη-μέλη να πατάξουν την διαφορά όταν δεν το κάνει το Κοινοβούλιο στον οίκο του. Ευχαριστώ πολύ Κυρία Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, πρώτα απ' όλα ε, να πω στο λίγο χρόνο που έχω στη διάθεσή μου ότι θα ήθελα να μιλήσω για την πολιτική διαφθορά και την απάτη. Ε, λυπούμε που σε αυτήν την ε, έκθεση ασχολούμαστε μονάχα με άλλου ε, είδους απατών, ενώ το Κοινοβούλιο αντιμετωπίζει τούτη τη στιγμή συγκεκριμένη διαφθορά και απάτη τριών μελών του ε, βουλευτών. Βεβαίως έχω την εντύπωση κιόλας ότι αυτοί οι τρεις βουλευτές είναι μονάχα η κορυφή του παγόβουνου, γιατί γίνονται τόσοι πολλοί διαγωνισμοί, γίνονται τόσες πολλές διαδικασίες που προϋποθέτουν ε, ε, πόρους και χρήση πόρων που πραγματικά πρέπει να πούμε ότι πάνω από το 50% ε, της τάξης των πολιτικών είναι διεφθαρμένη και από, την πλευρά μας και από την πλευρά των πολιτών βλέπουμε ότι δεν υπάρχει πια αγωνιστικότητα δηλαδή όλοι παραδέχονται την κατάσταση και απλώς συμφωνούν και λένε δεν βαριέσαι τι να κάνουμε και μετά κλείνουν σχολεία και δημιουργούνται προβλήματα. Ευχαριστώ. Μιλητών, η κυρία Γκράσλε για δύο λεπτά θα πάρει το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητέ Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Η έκθεση για το 2009 φέρνει πολλές καινοτομίε. Για πρώτη φορά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να ταξινομήσει το ύψος των απατών και ε, παρατυπιών. Δυστυχώς το πρόβλημα ακόμα ε, δεν το έχουμε αντιμετωπίσει και προσπαθείτε να το ωρεοποιήσετε. Κύριε Επίτροπε, δεν μου άρεσε καθόλου αυτό με στατιστικές μεθόδους. Άλλη καινοτομία. Το σύστημα EMS, ε, διαχείρισης ε, παρατυπιών. Σε 800 σημεία συλλέγονται στοιχεία στατιστικά και όχι σε 50 όπως ήταν μέχρι τώρα. Άρα αυξάνονται οι παρατυπίες 43% στην Γεωργία 23% στα διαρθρωτικά και σύνολο φτάνει μέχρι και 109%. Με οδύνη βλέπουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει πολύ μεγάλη υπομονή με τα κράτη-μέλη στην εφαρμογή, γιατί η εφαρμογή χωλαίνει, ε, σέρνεται και το λέει πολύ καλά η έκθεση αυτό. Γι' αυτό ζητάμε πλήρως να εφαρμοστεί το σύστημα EMS και ε, μόνο όταν θα λειτουργεί καλά και θα έχουμε αξιόπιστα στοιχεία θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την απάτη και τις παρατυπίες. Μας ανησυχεί η κατάσταση στην Ιταλία. Πρωταθλητής με μεγάλη διαφορά στην απάτη. 60% ε, των απατών και των υποψιών πέφτουν στην Ιταλία. Ε, άρα θα πρέπει να υπάρξει ένα πρόγραμμα ε, δράσης με ειδικά μέτρα για να βοηθήσουμε την Ιταλία. Ευχαριστώ πολύ την Όλαφ και τους υπαλλήλους της ε, γιατί ε, πραγματικά αξιόλογη δουλειά που κάνουμε. Εμείς σας υποστηρίζουμε και θέλουμε να τις υποστηρίξει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για ποιο λόγο υπάρχει πρόβλημα στην πρόσβαση ε, στην Τράπεζα Δεδομένων. Αν θέλει, υποτίθεται ότι θέλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δουλεύει όλα και το, θεωρείτε θεωρείται σημαντικό. Περιμένουμε απαντήσεις. Ευχαριστώ. κυρία Η κυρία Φλασίκοβα για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και να υποστηρίξω τον εισηγητή στην κριτική ε, που ασκεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την έκθεσή της. Γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εμένει στα στοιχεία που διαβιβάζουν τα κράτη-μέλη. Δεν αρκεί αυτό, κύριε Επίτροπε. Θα πρέπει να εφαρμόζεται τις ε, νεότερες ε, και πιο σύγχρονες μεθόδους για τη συλλογή ε, στατιστικών στοιχείων για να μην πλανώνει διάφορες σκιές και υποψίες σε πολλές καταστάσεις. Παράδειγμα, ορισμένα κράτη-μέλη που παίρνουν πολλά κονδύλια εμφανίζουν χαμηλό ποσοστό απατών. Αυτό είναι πραγματικό ή στατιστικό στοιχείο. Μήπως δεν συλλέγουν αρκετά στοιχεία, γι' αυτό δεν βρίσκουν απάτες. Προσπαθεί να μας πείσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι μπορούμε ε, να βάλουμε ποσοστώσεις του επιτρεπτού σφάλματος. Ε, E, zgadzam się z panem sprawozdawcą, że... Θα ήθελα να πω δεν θα πρέπει εδώ πέρα δεν θα πρέπει να πω εδώ πως θα πρέπει τις, τις παρατυπίες με την απάτη δεν θα πρέπει να τις αναμειγνύουμε. Και έχουμε και μερικές οριακές παρατυπίες. Τώρα για τα όσα υπόθηκαν για την έκθεση που μας υποβάλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα με βρείτε σύμφωνο. Είναι πολύ λίγες οι πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας για τη διάσταση της απάτης. Νομίζω πρέπει να δούμε το θέμα σε μεγαλύτερο βάθος, με περισσότερες λεπτομέρειες και θα ήταν καλύτερο να μας έχετε δώσει πιο συγκεκριμένες πληροφορίες. Αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να δώσουμε τη μάχη κατά της διαφθοράς με όλα τα όπλα που έχουμε στη διάθεσή μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα πρέπει τα κριτήρια που ακολουθούμε να εξασφαλίζουν τη διαφάνεια, να μην υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων και να εξασφαλίσουμε επίσης την ε, μέγιστη ευκρίνεια στη χρήση των ευρωπαϊκών κονδυλίων με συστηματικούς ελέγχους. Ευχαριστώ. για ένα λεπτό επίσης. Πρόεδρε, χαίρομαι για την έκθεση, αλλά για θλιβερό λόγο γιατί διαπιστώνουμε η απάτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παραθέτω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπαίνει σε λεπτομέρειες για την απάτη και οι παρατυπίες εξετάζονται πολύ γενικά. Και συνεχίζεται ε, η απάτη. Στη Πολωνία, Ρουμανία και Βουλγαρία αυξάνεται μάλιστα. Η Ισπανία, η Ιταλία είναι ε, υπεύθυνε για τις περισσότερες παρατυπίες και τα τελευταία χρόνια μόλις 10% ανακτήθηκαν πραγματικά από τα κονδύλια που ζητούσαμε και χώρες που έχουν λάβει ε, ειδική ενίσχυση για να μπουν στην Ένωση για τη Γεωργία και την Ήπεθρο. Όλα αυτά τα λέει η έκθεση. Μπράβο που τα γράφει. Πολύ καλό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως τι θα κάνει για να το αντιμετωπίσει. Για πόσο καιρό ακόμα θα ανεχόμαστε την απάτη και πόσο καιρό ακόμα θα πληρώνει τα σπασμένα ο πολίτης. Σε ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Ματσόνη τώρα για δύο λεπτά. Ε, ε, Θέλει να κάνει ε, μια ερώτηση στον κύριο Χάρτογκ. For, Mr. Ε? yes. Έχετε 30 δευτερόλεπτα σας παρακαλώ κύριε Στάς. Ναι, κύριε Χάρτογκ, άκουσα καλά την ομιλία σας, αλλά άκουσα και τον κύριο Γκάιερ που είπε κάποια στιγμή ότι δύο καθαρή συνεισφορείς, ε, το Ηνωμένο Βασίλειο και οι κάτω χώρες, υπολείπονται ε, κατά πολύ. Εσείς τι θα κάνετε που καταδικάζετε τα υπόλοιπα κράτη-μέλη για να φροντίζετε στη χώρα σας και η Ολλανδία ίδια να μην ε, παρατυπεί. Ο κύριος Χόρτοκ μπορεί να απαντήσει για 30 δευτερόλεπτα. Ευχαριστώ τον συνάδελφο για την ερώτηση. Αν διαβάσετε καλά την έκθεση θα διαπιστώσατε τα γεγονότα. Εγώ δεν μιλώ εξ ονόματος της ε, ε, Βρετανίας, αλλά το κάτω χωρών είναι τα χαμηλότερα, από τα χαμηλότερα ε, περιστατικά και όταν βρίσκουμε απάτη την πατάσουμε πρέπει να σας πω. Ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζουμε. Κυρία Ματσόνη για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι εκτιμούμε ιδιαίτερο στην εργασία του εισηγητού, η οποία όμως καταδεικνύει εν μέρη έλλειψη ε, προσοχής, ε, τουλάχιστον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο, γιατί πέρσι εμείς είχαμε σημειώσει προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάποιες ειδικέ δράσεις που θα έπρεπε να αναλάβει έτσι ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί σε αυτόν τον κεντρικό στόχο της προστασίας των οικονομικών συμφέροντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς επίσης και των πολιτών της Ευρώπης μέσω και των απατών και των παρατυπιών. Ε, σύμφωνα και με αυτά που λέει ο ε, εισηγητής, ε, δεν έχει μειωθεί η χρήση των ιδίων πόρων και επίσης οι καταγεγραμμένες παρατυπίες και απάτες ως ποσοστό είναι ακόμα πάρα πολύ υψηλέ Επίσης και σε όσον αφορά την ανάκτηση των πόρων πρέπει να πούμε ότι δυστυχώς δεν επιτύχαμε λαμβάνοντα υπόψη τα συγκεκριμένα στατιστικά στοιχεία. Στην έκθεση της περσινής χρονιάς είχε πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να παρέμβει σε ορισμένες κατηγορίες. Ε, και εγώ θα επικεντρωθώ σε τρεις κατηγορίες. Πρώτον, η ευαισθητοποίηση των κρατών μελών, κυρίως όσον αφορά ε, τους μηχανισμούς ε, κοινοποίησης και αναφορά των κρατών μελών. Δεύτερον, η σαφήνεια των κανονισμών. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να γίνει σαφής αναφορά στις παρατυπίες, τις απάτες και τα λάθη. Τρίτον, μόνο ασφαλή στοιχεία και συγκεκριμένα έτσι ώστε να μπορούμε ε, να προχωρήσουμε σε συγκεκριμένα συμπεράσματα αλλά βεβαίως ε, και να προβλεφθεί ε, η καταγραφή όλων των στοιχείων στο website με τρόπο απλό και κατανοητό. Επίσης πρέπει να, πρέπει να πω ότι η ελλειπής εναρμόνιση των εθνικών συστημάτων αφήνει παραθυράκια για παρατυπίες και απάτες. Επανειλημμένα Αναφέρθηκε το, η, Ιταλία. Η Ιταλία αναφέρεται άλλωστε ε, και στο έγγραφο του δικού μας συγητή. Να πω, αν μου επιτρέπετε, ότι ε, σίγουρα εμείς έχουμε εξαιρετικά βραδείς χρόνους πιστοποίησης ε, και η ποινική δικαιοσύνη αλλά και η διοίκηση προχωρούν με πάρα πολύ αργούς ρυθμούς. Αλλά εάν είχαμε όμως σαφείς ορισμούς για το τι είναι παρατυπία, τι είναι απάτη και τι είναι λάθος, τότε τα πράγματα θα ήταν πολύ πιο εύκολα. Ευχαριστώ και συγγνώμη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 Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα να συγχαρώ τον εισηγητή. Κατά την άποψή μου είναι πάρα πολύ σημαντική η δραστηριότητα αυτή και το Κοινοβούλιο και ε, το Ελεγκτικό Συνέδριο και τα Εθνικά Ελεγκτικά Συνέδρια και τα Εθνικά Κοινοβούλια πρέπει να συνεργάζονται έτσι ώστε να υπάρχει διαφάνεια. Ε, Βεβαίω ε, και η συνεργασία του Κοινοβουλίου είναι πάρα πολύ σημαντική. Νομίζω ότι όλοι εμείς θα πρέπει να μην έχουμε κανένα μελανό στοιχείο. Ε, θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ καθαροί απέναντι στου εαυτούς μας πρώτα έτσι ώστε ε, να μπορέσουμε να είμαστε εντάξει και προς τα έξω. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι εμείς ε, πρέπει να ξεχωρίσουμε τις παρατυπίες με τις απάτε. Παρατυπία και απάτη δεν είναι το ίδιο πράγμα. Η απάτη θα πρέπει οπωσδήποτε να ε, παταχθεί ενώ η παρατυπία ε, θα πρέπει ε, να αντιμετωπιστεί με τρόπον ώστε όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς να γνωρίζουν όσο γίνεται αναλυτικότερα και σαφέστερα τους κανόνες έτσι ώστε να μπορούν να τους εφαρμόζουν και, στην κατανομή, και υπάρχουν χώρες οι οποίες παρουσιάζουν μεγαλύτερα προβλήματα. Thank Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να συγχαρώ και την ε, σκιώδη εισηγήτρια και τον εισηγητή για τη δουλειά που κάνανε σε αυτή την έκθεση, γιατί οι φορολογούμενοι θέλουν να ξέρουν πώς γίνεται καλή χρήση των χρημάτων τους. Νομίζω πως η τελευταία ομιλήτρια το τόνισε. Η διαφορά μεταξύ παρατυπίας και απάτης είναι σημαντική, γιατί για το κοινό μας ε, απάτη είναι κάτι το οποίο γίνεται με... Ε, δόλο, ενώ σφάλματα παρατυπίες είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει κατά λάθο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν θα έπρεπε όλα αυτά να αποτελούν μία κατηγορία γιατί υπάρχει μία διαφορά μεταξύ τους για τη γεωργία η οποία αναφέρθηκε από κάποιους συναδέλφου. Είναι σημαντικό να είναι απόλυτα διάφανος ο τρόπος με τον οποίο γίνονται οι πληρωμές στην γεωργία και εκεί έχουμε κάνει τεράστια πρόοδο. Όσο όμως προχωράμε προς τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ, καλό θα είναι να συνεχίσουμε να φέρουμε αυτές τις βελτιώσεις. Ε, πρέπει να σας πω πως η 24 με βρίσκει ιδιαίτερα σύμφωνη όπου μιλάμε για συστήματα ελέγχου. Ξέρω πως τα κράτη, το μέλος το οποίο εκπρόσωπο οι παραγωγοί έχουν νέους χάρτες στους οποίους πρέπει να δηλώσουν και ξέρετε πως έχει χρειαστεί πολλούς χρόνους και υπομονή για να κλείσει αυτό το έργο και ξέρω πως καμιά φορά τα άτομα παγιδεύονται από το σύστημα ενώ οι μεγάλοι παίκτες που μπορεί ενδεχομένως να και πιο ένοχοι σε κάποια απάτη είναι πολύ πιο δύσκολο να βρεθούν οπότε ε, θα πρέπει να προσέξουμε να μην τρομοκρατούμε τα μεμονωμένα άτομα. Γίνες, ο κύριος Μπαλτζούτης για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Ιβαν για την εκπόνηση της έκθεσης αυτής. Τα χρήματα των Ευρωπαίων φορολογουμένων θα πρέπει να πιάνουν τρόπο και να, τόπο συγγνώμη, και να αποδίδουν. Τα κράτη-μέλη να έχουν σωστούς ενεκτικούς μηχανισμούς για να ε, μπορούν να ανοιχνεύουν τις απάτες είναι πολύ σημαντικό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Όλαφ να συλλέγουν και να δέχονται στοιχεία αξιόπιστα και επίσης η ανάκτηση των ποσών πολύ χαμηλή και θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να παίρνουμε πίσω τα κονδύλια που δεν δικαιούνται όσοι τα χρησιμοποιούν. Επίσης, η έκθεση του Κοινοβουλίου και η αιτήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Προστασία των Οικονομικών Συμφερόντων της Ένωσης θα πρέπει να ε, την χάνουν ε, μεταχείριση και να δίνεται συνέχεια στα κράτη-μέλη και στο Συμβούλιο. Σα ε, παρακαλώ για δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Δυστυχώ η έκθεση αυτή για μια φορά ακόμα φέρνει τη διαπίστωση πώ πολλές επιδοτήσεις χρησιμοποιήθηκαν με σφαλμένο τρόπο και δεν ανακτήθηκαν έγκαιρα. Είναι λοιπόν ατελείς οι προσπάθειες που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να εξασφαλίσει στα κράτη-μέλη πως το ποσοστό σφάλματος θα είναι χαμηλού. Πολλοί συνάδελφοι είπαν πως θα πρέπει να δούμε τι σημαίνει παρατυπία και τι σημαίνει απάτη γιατί δεν γίνεται μια σαφής διάκριση. Νομίζω πως η προσέγγιση ε, συμπερίληψης κάποιων πράξεων στην παρατυπία είναι υπερβολικά γενικόλογη. Θα πρέπει να δούμε ποιες διαδικασίες παρατυπίας ε, συμπεριλαμβάνονται. Για την γεωργία το 85% των πληρωμών υποτίθεται ότι γίνεται κανονικά. Παρόλα αυτά σε κάποια κράτη-μέλη ο ρυθμός παρατυπιών είναι εξαιρετικά μεγάλος. Το σύστημα ανείχνευσης πολλές φορές δεν είναι αποτελεσματικό και δεν μπορεί κανείς να το θεωρήσει αξιόπιστο. Πιστεύω πως οι έλεγχοι θα γίνουν πιο αποδοτικοί αν έχουμε πιο συγκεκριμένα στοιχεία στα χέρια μας για να εξασφαλίσουμε πως τα εθνικά όργανα δίωξης απάτης και παρατυπιών θα είναι πιο αποδοτικά. Αυτές οι παρατυπίες θα πρέπει να ξεπεραστούν και να βελτιωθούν τα συστήματα που οδηγούν σε αυτές. Για το ελεγκτικό συνέργεια αναφέρεται σε 30% περίπου ποσοστό παρατυπίας από τα αρμόδια εθνικά όργανα. Άρα λοιπόν τα κράτη-μέλη θα πρέπει και αυτά να δουν τι μπορούν να κάνουν για να βελτιώσουν τους μηχανισμούς παρακολούθησης, ανείχνευσης και διόρθωσης. Ζητώ λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βρει περισσότερες προφορίες για τα συστήματα που λειτουργούν στα κράτη-μέλη και να μας πει και ποια μέτρα θα ήταν τα κατάλληλα για να ξεπεράσουμε παρατυπίες και δυσλειτουργίες. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Καταλίνη για αυτή την προσπάθεια που έκανε. Με ιδιαίτερη σοβαρότητα κατάφερε να φέρει σε πέρας ένα θέμα το οποίο είναι εξαιρετικά επίμαχο και είναι η προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Θα ήθελα να τον συγχαρώ γιατί πρέπει να δούμε ποια ορολογία θα χρησιμοποιούμε απάτη. Απάτη πάντοτε ε, κρύβει την έννοια του δόλου και της παρατυπίας από την άλλη μεριά. Δεν θα πρέπει να τα αναμειγνύουμε έτσι ώστε να καταλήγουμε σε ποσοστά τα οποία είναι εντυπωσιακά. Τώρα για τις προθεσμίες και τις καθυστερήσεις που έχουμε στην αποκάλυψη αυτών των σφαλμάτων, παρατυπιών κτλ. που οδηγούν σε δύσκολη θέση τα κράτη-μέλη. Να σας πω πως μιλάμε για προθεσμίες οι οποίες αργούν να δώσουν τελικά στοιχεία. Αυτή τη στιγμή ο μόνος ε, ε κύκλος που έχει κλείσει είναι αυτός που είναι το, λίγη το 1999. Αυτή τη στιγμή ε, ερευνώνται οι υποθέσεις από το 2000 μέχρι το 2006. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια σημαντική καθυστέρηση. Θα πρέπει όλα αυτά τα ζητήματα να τα δούμε στα πλαίσια του κώδικα διοντολογίας και να δούμε και το θέμα της Κίνας και των τρίτων χωρών. Έχουμε ξεφύγει από τον χρόνο. Ο κύριος Κοντζολίνο για ένα λεπτό. Ένα λεπτό ακριβώς παρακαλώ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή γιατί όλα αυτά τα στοιχεία είναι πάρα πολύ σημαντικά και θα πρέπει βεβαίως να προσαρμοζόμαστε στα νέα ε, δεδομένα ελέγχου και εδώ προκύπτει ένα ζήτημα κυρίως όσον αφορά την αναφορά των κρατών σχετικά με τις παρατυπίες και τις απάτες. Βλέπουμε ότι υπάρχουν χώρες οι οποίες συστηματικά ανακοινώνουν και διαβάζουν πολύ χαμηλά ποσοστά παρατυπίας και απάτης και νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρξει σαφήνεια όσον αφορά τα στατιστικά στοιχεία τα οποία μεταδίδονται. Επίσης ε, ε, πρέπει να διαπιστώσουμε ότι το σύστημα ανάκτησης ε, δεν είναι αποτελεσματικό. Όμως βλέπουμε ότι υπάρχει μια καλή τάση μακροχρόνια Δηλαδή ε, δεν είναι ε, δυνατόν να πούμε ότι ε, τα κράτη-μέλη συνεργάζονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση με τον τρόπο και στο βαθμό που θα έπρεπε. Επομένως πιστεύω ότι θα πρέπει να τροποποιηθεί ο κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις δημόσιες αναθέσεις και να υπάρχει κατάλογος αυτών που λαμβάνουν χρήματα ευρωπαϊκά. Ένα λεπτό επίσης. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε θα ήθελα να συγχαρώ και εγώ τον εισηγητή για την εξαιρετική δουλειά του στην ετήσια έκθεση για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων τη Ευρωπαϊκή Ένωση, όπω και την καταπολέμηση τη απάτη η έκθεση καλύπτει διεξοδικά όλου του τομεί όπου τα κράτη μέλη εκτελούν τον προπολογισμό όπω γεωργία συνοχή προνταξιακά ταμεία και τη συλλογή των ιδίων πόρων τη ευρωπαϊκή ένωση μέσω των τελωνιακών δασμών. συμφωνώ απόλυτα ότι είναι απαραίτητη η βελτίωση τη εποπτείας των προενταξιακών κονδυλίων δεδομένη τη εμπειρία του 2009, όπω και ότι είναι απαραίτητη η συνεχή παρακολούθηση του έργου τη Όλαφ και όχι μόνο όταν συζητείται ετήσια έκθεση. θα ήθελα τέλο κύριε πρόεδρε να τονίσω ότι η έκθεση μα προσφέρει σημαντικά ευρήματα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στις συζητήσεις που έχουν ξεκινήσει τόσο για την αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού όσο και για το σχεδιασμό της πολιτικής συνοχής μετά το. 2013. Πολύ συνεπής και στον χρόνο. Ο κύριος Κάλφιν πιστεύω να σας ακολουθήσει. Ένα λεπτό παρακαλώ. much, uh, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, ε, θα μιλήσω βουλγαρικά. Λοιπόν, θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή ε, για τη μεθοδικότητα στο έργο του. Επανειλημμένα έχουμε αποδείξει ότι το Κοινοβούλιο φροντίζει να γίνεται χρηστή διαχείριση των κοινοτικών πόρων και των χρημάτων των φορολογουμένων. Θα ήθελα να καλύψω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να θεσπίσει κανόνες πολύ πιο σαφείς και πολύ πιο ε, διάφανους. Δεν κάνει διάκριση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανάμεσα στην απάτη, ε, στα σφάλματα και εισάγει μάλιστα και τον όρο υποψία που έρχεται να θολώσει ακόμα περισσότερο το τοπίο. Θα παρακαλούσα οι κανόνες να είναι πιο σαφείς και πιο ε, καλή η πληροφόρηση από τα κράτη-μέλη και οι εθνικές δηλώσεις. Είσαι ακριβή στον χρόνο. Τώρα ερχόμαστε στο Catch the Eye. Έχουν ζητήσει το λόγο τρεις συνάδελφοι. Η κυρία Μπασέσκου καταρχάς. Ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. πολλά κονδύλια ευρωπαϊκά δεν χρησιμοποιούνται για τον λόγο για τον οποίο έχουν δοθεί και επίσης ε, η δυσκολία ανάκτησης ε, είναι σαφής. Ε, το έχω ξαναπεί και πρέπει να το ξαναπώ. Έχουμε δυνατότητα και έχουμε περιθώριο μείωσης της διαφθοράς στους δημόσιους διαγωνισμούς μέσω τροποποίησης του κανονισμού. Ε, η Ρουμανία έχει μεγάλες δυσκολίες ε, όσον αφορά την ε, μείωση των παρανόμων δραστηριοτήτων, όπως και άλλες χώρες άλλωστε. Πάντως πρέπει να πούμε ότι τους τελευταίους μήνες έχουν, έχουν υπάρξει στη χώρα πάρα πολύ έλεγχοι, καθώς επίσης και επιδρομές των διοκτικών αρχών, έτσι ώστε να ε, διασφαλιστούν τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης. Αναφέρομαι κυρίως στο λαθρεμπόριο τσιγάρων. Ο κύριος Όμπερ παρακαλώ, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τα λάθη γίνονται ε, από απροσεξία ή από άγνοια. Η απάτη όμως όχι. Προϋποθέτει δόλο. και ε, Καμιά φορά ε, όποιος διασπαθίζει δημόσια κονδύλια ε, σήμερα θεωρείται ρομπέν των δασών και όχι απατεώνας. Μα τα χρήματα αυτά είναι των φορολογουμένων. Χρειάζονται υψηλά πρόστιμα χρηματικά αλλά και άλλα μέτρα. Περισσότερη διαφάνεια, σαφής διαχωρισμός των ορισμών, τι εστί παρατυπία, τα σταλία, απάτη και τι σφάλμα. Δεν μπορεί ο ένας να ρίχνει ο βάρος των άλλων ή να εμποδίζει όλη αυτή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κτλ. Χρειάζεται δράση οπωσδήποτε για να μπει τάξη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Και ο κύριος Πίπερ για ένα λεπτό παρακαλώ θα πάρει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η απάτη στις επιδοτήσεις και τα ασταλίες ε, στα κοινοτικά κονδύλια μπορεί να έχουν μειωθεί το τελευταίο διάστημα, αλλά ο κόσμος παραμένει επικριτικός. Και σωστά. Πολλοί θεωρούν ότι ε, δεν ανακτούμε σωστά ε, τα ποσά που έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως και η ζημία είναι για όλους τους φορολογούμενους πολίτες. Και θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, να αντιδράσει την κατάσταση αυτή, μπορώ να σας πω να δώσει και λιγότερα του χρόνου στα κράτη-μέλη μέχρι να ανακτηθούν τα κονδύλια που πρέπει. Επίσης, σε περίπτωση που δεν έχουμε σχεδόν καθόλου παρατυπίες, θα πρέπει να καταλαβαίνουμε ότι όποιο δεν δηλώνει τι παρατυπίε δεν θα πρέπει να φροντίσει να επιστραφούν τα ποσά και κρατάει τα χρήματα. Η Ισπανία, η Γαλλία και άλλε χώρε καλούνται στην έκθεση να ανοίξουν τα χαρτιά του. Και παρακαλώ να ενισχυθούν οι έλεγχοι από την Επιτροπή. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ πολύ κύριε Πίπερ. Κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, εδώ τελειώσαμε και τη διαδικασία Catch the Eye. Το λόγο θα πάρει ο Επίτροπο ο κύριο Σεμέτα. Mr. Commissioner. Uh, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα για μία ακόμα φορά να ευχαριστήσω τον κύριο Ήβαν ε, για την επικοδομητική του συνεισφορά στην ε, συζήτηση μέσω της εξαίρετης έκθεσης καθώς επίσης ε, και που αποτέλεσε βάση καλή για αυτήν την συζήτηση που έλαβε χώρα σήμερα και που ακολούθησε την έκθεση Επιτροπής για το 2010. Βεβαίως ε, θα βελτιωθεί το περιεχόμενο του 325 λαμβάνοντα υπόψη ε, τις ε, προτάσεις οι οποίες αναφέρθηκαν στη διάρκεια της συζήτησης και βεβαίως είναι γεγονός ότι πρέπει να βελτιωθούν οι στατιστικές, έχουν ήδη βελτιωθεί, αλλά πάντα υπάρχει δυνατότητα περαιτέρω βελτιώσεως και γι' αυτό λοιπόν εμεί θα ζητήσουμε τα κράτη-μέλη να μας υποβάλουν περισσότερες πληροφορίες, καθώς επίσης ε, να κάνουν καλύτερο διαχωρισμό ανάμεσα στις παρατυπίες ε, και τι απάτε, καθώ επίση και να δίνουν σαφείς ε, πληροφορίε και για τι παρατυπίες και για τι απάτε. Έχετε δίκιο κυρία Γκρέσλερ ότι μπορούμε να κάνουμε βελτιώσεις στο σύστημα ε, διαχείρισης ε, των ε, παρατυπιών. Επίσης το θέμα της διαφάνειας όσον αφορά το ποιοι είναι οι αποδέκτες των χρημάτων. Είναι αλήθεια ότι πρέπει να υπάρχει σαφής ε, κατάλογος των δικαιούχων και αυτή είναι πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επίσης η Επιτροπή συμμερίζεται την άποψη ότι τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί από τα κράτη-μέλη για την καταπολέμηση της απάτης και της διαφθοράς ε, έχουν κάνει το σύστημα πιο αποτελεσματικό αλλά και εδώ υπάρχει δυνατότητα και περιθώριο για περαιτέρω βελτίωση. Ε, ε, σχετικά με τα λεγόμενα του κυρίου Γκάγερ πρέπει να πω ότι ναι όντως η απάτη δεν γνωρίζει εθνικά σύνορα και δεν είναι πρόβλημα για τα μεν κράτη-μέλη και όχι για τα δε και δεν αφορά μονάχα τις νέες χώρες μέλη αλλά αφορά και τις ε, παλαιότερες χώρες μεταξύ των οποίων και τις χώρες τις οποίες εσείς ονομάσατε ή στην ε, ε, παρέμβασή σας και βεβαίως θα πρέπει τα ζητήματα αυτά ε, να ε, αντιμετωπιστούν σωστά σε όλες τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρέπει να πω ότι και εγώ ίδιος αλλά και οι υπηρεσίες μου έχουμε δεσμευτεί στην βελτίωση της ε, κατάστασης ε, και η έκθεση για το 2010 θα είναι οπωσδήποτε ε, πολύ υψηλής ποιότητος. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε, λέει η Πρόεδρος. Ο εισηγητής ο κύριος Σίβα. Έχετε το λόγο κύριε Σιγητά για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ και εγώ τον Επίτροπο και όλους τους συναδέλφους που συνεισέφερα ε, στην εκπόνηση της έκθεσης με τροπολογίες ή με τη σημερινή τους τοποθέτηση. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τους και ηγητές με τους οποίους είχα άριστη συνεργασία. Η έκθεση αυτή είναι ο καρπός της καλής μας συνεργασίας. Θα ήθελα και πάλι να πω ότι αυτό που χρειάζεται είναι ακριβώς αφής διαχωρισμός του ορισμούς μεταξύ παρατυπιών και απάτης. Μπορούμε να δεχθούμε κάποιο σφάλμα, ε, να έχουμε κάποια ανοχή στις παρατυπίες, αλλά μηδενική ανοχή στην απάτη. Χρειάζεται η εθνική δήλωση διαχείριση να υπογράφεται από ένα πολιτικό πρόσωπο, από το πολιτικό προϊστάμενο, τον Υπουργό. Προσβλέπουμε ε, στον έλεγχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την απλουστευμένη διαδικασία, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να διαχειριζόμαστε με σωστό τρόπο ε, τους πόρους του προπολογισμού. Σε ό,τι αφορά τους διαγωνισμούς και ε, την εκτέλεση του προϋπολογισμού, Ξέρουμε ότι σε πάρα πολλές χώρες είναι υπερβολική η γραφειοκρατία, η οποία έχει ως στόχο μεν την καταπολέμηση της απάτης, αλλά ταυτόχρονα ε, δημιουργεί και τις προϋποθέσεις για απάτη ε, στη διαχείριση των κοινοτικών κονδυλίων. Και διαφθορά. Γιατί πολλές φορές τα χρήματα αυτά καταλήγουν σε χέρια πολιτικών. Όταν έχουμε λοιπόν υποψίες ε, για απάτη μπορούμε να φτάνουμε και μέχρι διακοπή ή αναστολή των πληρωμών και των εκταμιεύσεων. Ευχαριστώ. Εδώ κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο στις 12. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα έλθουμε στην ώρα των ερωτήσεων στη συνέχεια.